Right, uh, Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι τρεις και εννέα λεπτά. Γι' αυτό και κυρίσω την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης και σας καλωσορίζω. Πρώτο σημείο, έγκριση της σημερινής διάταξης. Αν δεν υπάρχουν σχόλια, εγκρίνεται. Σημείο 2, ανακοινώσεις του Προέδρου. Δεν έχω καμία ανακοίνωση επί του παρόντος. Οπότε περνάμε στο σημείο 3. Έγκριση των πρακτικών της προηγούμενης συνεδριασής μας. Αν δεν υπάρχουν ε, σχόλια για τα πρακτικά της συνεδριάσεως 13 Φεβρουαρίου, μέχρι αύριο θεωρούνται εγκεκριμένα. Σημείο 4. Προηγουμένως όμως θέλω να καλωσορίσω εδώ έναν ιδιαίτερο προσκεκλημένο που κάλεσε εδώ, τον ε, συνάντησα βέβαια πριν στην αίθουσα του πρωτοκόλλου, πάντως να ξέρετε είναι μεγάλη τιμή για μας που μπορούμε να έχουμε μαζί μας στη συνεδρίασή μας σήμερα τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου της Αιθιοπίας, τον κύριο Αμπαντούλα και Καλώς ήρθατε. Τον συνοδεύει ο πρόεδρος της Επιτροπής του Κοινοβουλίου Εξωτερικές Υποθέσεις, ο κύριος Βακάουλ. Καλώς ήρθατε. Είναι μια σημαντική χώρα με την οποία συνεργαζόμαστε η Αιθιοπία και είναι εδώ για την ε, μεικτή συνέλευση, οπότε πολύ χαίρομαι που τον έχουμε μαζί μας και θα δει πώς δουλεύουμε στην ΑΦΕΤ. Και τώρα περνάμε στο σημείο 4. Συνέπειες και εφαρμογή της απόφασης του Δικαστηρίου τη Ευρωπαϊκή Ένωση στην υπόθεση Συμβούλιο κατά του μετόπου Πολυσάριου όσον αφορά τι εμπορικέ σχέσει και τη συνεργασία τη Ευρωπαϊκή Ένωση με το Μαρόκο. Καλωσορίζω λοιπόν εδώ του συναδέλφου από την Επιτροπή Ίντα γιατί μαζί του θα συνεδριάσουμε εδώ. Θέλω εδώ πέρα να καλωσορίσω τον κύριο Γιώστο Κότερ που είναι αναπληρωτή στη Γενική Διεύθυνση Trade, τον κύριο Αντώνη Κασταλδιανάκη που είναι διευθυντής για την ασφάλεια και τη διευκόλυνση εμπορίου, τη διεθνή συνεργασία στην Γενική Διεύθυνση Ταξούντ. Πολύ Χαίρομαι λοιπόν που θα συζητήσουμε εδώ θέματα συνεργασίας, θέματα ε, καταπολέμησης της τρομοκρατίας κτλ. Η εταιρική σχέση που έχουμε με το Πολυσάριο βέβαια εμπίπτει στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου. Ο κύριος Πίκια θα μας ενημερώσει για το τι έχει γίνει μέχρι τώρα, θα μας ε, πει επίσης πώς θα προχωρήσουμε και ο κύριος ε, Λάνκε θα εισάγει το θέμα του κ. Καστιγιανάκη, ο οποίος θα μας μιλήσει για το εμπόριο και την ελευθέρωση αγροτικών προϊόντων. Η συνάντηση αυτή θα είναι μια καλή ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις μαζί για τις σχέσεις μας με το Μαρόκο. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Α, είσαστε εκεί. Παρακαλώ. Γιατί δεν είσαστε εδώ. Καλά. Εντάξει, δεν πειράζει. Θα μείνετε εκεί. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρόεδρε, πολύ χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ και όντως και η ΑΦΕΤ και η ΙΝΤΑ βρίσκονται εδώ. Χαίρομαι που είναι εδώ και οι δύο αυτές επιτροπές, αλλά και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης επίσης, όπως επίσης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εδώ, στο ίδιο έδρανο λίγο πολύ, παρόλο που συνήθως κάθονται χωριστά. Λοιπόν, ευχαριστούμε για την πρόσκληση πρώτα απ' όλα. Και αρχίζω Αναφερόμενος στην ενημέρωση που δόθηκε στην Επιτροπή ΑΦΕΤ πριν από λίγο καιρό, ήταν αρχές Ιανουαρίου, από την Ευρωπαϊκή Πίεση Εξωτερικής Δράσης αμέσως μετά από την απόφαση του δικαστηρίου. Θέλω να υπενθυμίσω ποια είναι η βάση της απόφασης αυτής. Στις 21 Δεκεμβρίου το δικαστήριο αποφάσισε για την προσφυγή όσον αφορά το γενικό πλαίσιο της συμφωνίας για τα αγροτικά προϊόντα. Ε, ανεστάλλει η απόφαση και ανετράπει η προηγούμενη απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου για την ίδια αυτή συμφωνία του 2015. Ως αποτέλεσμα, η γεωργική συμφωνία, η απόφαση δηλαδή του Συμβουλίου παραμένει έγκυρη όσον αφορά την εφαρμογή της συμφωνίας. Τώρα υπάρχουν σημεία στη συμφωνία αυτή που δεν καλύπτουν ρητά την ε, περιοχή της Δυτικής ε, Σαχάρας και όντως δεν την καλύπτουν. Αυτό είναι ένα πολύ ευαίσθητο, περίπλοκο θέμα με έναν βασικό εταίρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρίσκεται στα σύνορά της. Πρέπει φυσικά να σεβαστούμε την απόφαση, εννοείται, και πρέπει να το κάνουμε και με τέτοιο τρόπο ώστε να διατηρηθούν οι σχέσεις μας με το Μαρόκο, γιατί εδώ πέρα υπάρχουν σημαντικά πολιτικά συμφέροντα, οικονομικά συμφέροντα επίσης και φυσικά και χρειαζόμαστε και το Μαρόκο ως εταίρο για πολλά και διάφορα ζητήματα όπως είναι η ασφάλεια, η περιφερειακή σταθερότητα, η μετανάστευση και η αντιτρομοκρατία. Αναγνωρίζουμε ότι τον τελευταίο 1,5 χρόνο όσο ήταν σε κρεμότητα οι δικαστικές αποφάσεις είδαμε να μειώνονται οι δραστηριότητες ε, στα πλαίσια των σχέσεών μας με τον Μαρόκο εξαιτίας ακριβώς αυτής της δικαστικής διαμάχης αλλά και ε, του θέματος της κλιματικής αλλαγής. Τώρα μετά την απόφαση έχουμε κάθε συμφέρον να αποφύγουμε παρετέρω ταραχές όσον αφορά την σύγκρουση στην Δυτική Σαχάρα. Στόχος μας πρέπει να είναι να βοηθήσουμε την ειρνευτική διαδικασία του ΟΗΕ προκειμένου αυτή να συνεχιστεί. Ήμασταν σε επαφές με τις αρχές του Μαρόκο μετά την ανακοίνωση της απόφασης και αναγνωρίζουν ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί. Το θέμα δεν είναι το αν, το θέμα είναι το πώς θα γίνει αυτό. Και είναι επίσης πολύ σημαντικό για μας να αναλάβουμε και δράσεις οι οποίες από τη δικιά τους την ε, άποψη να μην δυσκολεύουν την πνευτική διαδικασία για τη Δυτική Σαχάρα. Ως Ευρωπαϊκή Ένωση Εννοείται ότι δεν πρέπει να καταδικάσουμε την θέση του Μαρόκο, ούτε τη θέση του Πολυσάριο, αλλά από τη στιγμή που οποιαδήποτε λύση απαιτεί στενή συνεργασία από το Μαρόκο και πολιτικής φύσεως αλλά και τεχνικής πρέπει να επιδείξουμε ευαισθησία στις απόψεις τους. Υπάρχει ευκαιρία λοιπόν τώρα για διάλογο. Το είπε και η Αντιπρόεδρος Μογκερίνη στη δήλωσή της, αλλά και ο υπουργό του Μαρόκο στις 21 Δεκεμβρίου. Πρέπει να χρησιμοποιούμε λοιπόν την δυνατότητα που έχουμε. Ο χρόνος βέβαια πιέζει. Πρώτα απ' όλα γιατί χώρες μέλη ε, περιμένουν από εμά να δράσουμε. Δεύτερον, υπάρχει πίεση και από την πραγματική οικονομία. Οι οικονομικοί φορείς πρέπει να γνωρίζουν που βρίσκονται. Έχουμε εκθέσεις που μιλούν για την ε, σημερινή νομική κατάσταση και δεν πρόκειται μόνο για τη Δυτική Σαχάρα, αλλά γενικότερα με το Μαρόκο. Επηρεάζονται δηλαδή από την απόφαση αυτή πολλές ε, επιχειρήσεις και στο Μαρόκο, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και άρα η ίδια η ζωή των πολιτών επηρεάζεται. Πρέπει επίσης να έχουμε υπόψη μας ότι υπάρχουν άλλες δύο δικαστικές υποθέσεις οι οποίες εκκρεμούν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για άλλες διμερείς συμφωνίες που έχουμε με το Μαρόκο. Αυτό στην πράξη για μας σημαίνει ότι η λύση που σχεδιάζουμε για την Αγροτική Συμφωνία, όσο και αν είναι δύσκολο, θα πρέπει να προκαταλάβει και οποιαδήποτε απόφαση έχουμε από το δικαστήριο και για τις άλλες δύο περιπτώσεις. Όπως είπαμε, είχαμε προκαταρτικές επαφές με το Μαρόκο τους τελευταίους δύο μήνες σε τεχνικό επίπεδο, αλλά υπήρξε και επίσκεψη από τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών του Μαρόκο που πήγε να δει την υπατή εκπρόσωπο. Οι επαφές έδειξαν ότι και οι δύο πλευρές αναγνωρίζουν ότι πρέπει να σεβαστούμε τη δικαστική απόφαση. Και οι δύο πλευρές συμφώνησαν για την σημασία που έχει η διατήρηση των σχέσεων και οι δύο πλευρές επίσης επιθυμούν να παραμείνει το παραδοσιακό εμπόριο που έχουμε με την Δυτική Σαχάρα, ανάμεσα στη Δυτική Σαχάρα και την Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή, και να υπάρξει συνέχεια, να αποφύγουμε προβλήματα στο εμπόριο τα οποία δεν είναι προς το συμφέρον κανενός. Σε σχέση τώρα με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, προσπαθούμε να δούμε πώς θα διορθωθεί η κατάσταση βάσει των όσων είπε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ότι δεν ήταν ε, σωστό έλειπε μια σωστή νομική βάση προκειμένου να εφαρμοστούν ε, προτιμησιακοί τελωνιακοί δεσμοί για εμπορεύματα που έρχονται από τη Δυτική Σαχάρα. Οπότε θα υπάρξει μια τροποποίηση στην ε, εμπορική συμφωνία. Για να το πετύχουμε αυτό φυσικά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας την ε, αιτιολόγηση που παρουσιάζει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Πρώτον, τα κριτήρια τα οποία αναφέρονται, δηλαδή τον καλύτερο δηλαδή, τρόπο να διασφαλιστούν διαβουλεύσεις με τους ενδιαφερόμενους και ο καλύτερος τρόπος είναι να φροντίσουμε τα μέτρα να είναι προς όφελος του κόσμου. Επίσης να φροντίσουμε τα μέτρα να είναι βιώσιμα όσον αφορά δηλαδή τις επιπτώσεις του στο περιβάλλον, να προστατεύει το περιβάλλον. Δεύτερον, οποιαδήποτε λύση θα πρέπει να σέβεται φυσικά τη δικαστική απόφαση, αλλά επίσης το διεθνές δίκαιο και τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη Δυτική Σαχάρα. Οποιαδήποτε λύση θα πρέπει να είναι συμβατή επίσης με την ειρηνευτική διαδικασία και δεν θα πρέπει να προκαταλαμβάνει το αποτέλεσμα της διαδικασίας και θα πρέπει αν γίνεται, να βοηθήσει στην ολοκλήρωση της διαδικασίας. Οπότε, εν κατακλείδη, μετά την απόφαση αυτή, θέλουμε να βρούμε την κατάλληλη νομική βάση όσον αφορά τις ε, προτιμησιακές ε, τελωνιακές ε, σχέσεις, να διατηρηθεί η παράδοση που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια και να μην πληγεί το εμπόριο με τη Δυτική Σαχάρα τη συνέπεια νομικού κενού που μπορεί να προκύψει. Αν τα καταφέρουμε, αυτό θα ήταν προς όφελος του πληθυσμού της Δυτικής Σαχάρας, αλλά και προς το συμφέρον των εμπορικών σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης Μαρόκο, που βέβαια έχουν κάπως αυλωθεί τα τελευταία χρόνια. Τέλος, και αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό, η προσέγγιση μας είναι συμβατή με την νευτική διαδικασία του ΟΙΕ. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ κύριε Πικέτ. Μας παρουσιάσατε και μας εξηγήσατε πράγματι την απόφαση του δικαστηρίου. Και μας είπατε για τις αδικές σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Μαρόκο. Από τη δικιά μας την Επιτροπή, αυτό που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, είναι να ακούσουμε κάποιες συμβουλές για το πώς θα προχωρήσουμε μετά την απόφαση αυτή. Τι σημαίνει στην πράξη η απόφαση αυτή. Να φροντίσουμε να μην υπάρχουν αρνητικές συνέπειες επί του εμπορίου. Εμπορίου ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Μαρόκο, αλλά και εμπορίου ανάμεσα στο Μαρόκο και τη Δυτική Σαχάρα. Όσον αφορά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, λοιπόν, δεν λέει ότι απαγορεύεται να μας έρχονται αγαθά από τη Δυτική Σαχάρα, αλλά ότι δεν μπορούν να εμπίπτουν στην κατηγορία των προτιμησιακών τελωνιακών δασμών. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν. Αυτή είναι η ερώτησή μου προς τον επόμενο μιλητή, που είναι αναπληρωτής διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Trade. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Πρόεδρε, να επανέλθω στο προηγούμενο σημείο που θίξατε για τις πολύ σημαντικές εμπορικές σχέσεις μεταξύ Βασιλείου του Μαρόκου και Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Έχω και μερικά νούμερα για να σας εξηγήσω καλύτερα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο πιο σημαντικός εμπορικός εταίρος του Μαρόκου. 55,7 του συνολικού εμπορίου για το 2016 και 27% από το Μαρόκο ήρθαν στην Ευρώπη, ενώ 52% των εισαγωγών του Μαρόκου ήταν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα πολύ σημαντική εμπορική σχέση με συνολική αξία αγαθό, αγαθών στα 34,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Και μιλώ μόνο για αγαθά. Εάν προσθέσετε σε αυτά και τις υπηρεσίες, έχετε άλλα 8,6 δισεκατομμύρια ευρώ για το 2015. Άρα και εντατική και σημαντική οικονομικά και πολιτικά σχέση, όπως εξήγησε και ο κ. Σαμπικέ, και εμπορικά βεβαίω. Το Μαρόκο έχει μάλιστα σημειώσει σημαντική πρόοδο στον τομέα της ρυθμιστικής προσέγγισης με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένας από τους λόγους για τους οποίους αποφασίστηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση το Μαρόκο να αποτελέσει την πρώτη χώρα με την οποία θα συνάψουμε DCFTA, δηλαδή σε βάθος συνολική ε, εμπορική συμφωνία. Ήδη άρχισαν οι εργασίες από το 2013 και τώρα έχουν προχωρήσει και βεβαίω και λόγω της αποφάσεως του δικαστηρίου αλλά και για άλλους λόγους οι διαπραγματεύσεις αυτές έχουν στην πραγματικότητα πάυσει, σταματήσει. Είναι σαφές ότι χωρίς λύση του νομικού προβλήματος που συζητούμε άλλωστε σήμερα το απόγευμα, θα είναι πολύ δύσκολο να επανακινήσουν οι ε, διαπραγματεύσει αυτέ. Και είναι προ συμφέρον και των δύο πλευρών, βεβαίω και τη Ευρωπαϊκή Ενώση από τη δική μα πλευρά και του Βασιλείου του Μαρόκου από την άλλη, να κάνουμε την απαραίτητη προσπάθεια για να το επιλύσουμε το πρόβλημα. Βεβαίω πάντοτε συμμορφούμενοι με την απόφαση του δικαστηρίου, κάτι το οποίο καθίστε απόλυτα σαφής και από τον εκπρόσωπο της, ε, Επιτροπή, της ε, Υπηρεσίας Εξωτερικών Δράσεων. Η απόφαση του δικαστηρίου του Δεκεμβρίου επιβεβαιώνει την νομιμότητα της αποφάσεως για την έγκριση της συμφωνίας με το Μαρόκο, της αποφάσεως του Συμβουλίου. Και αυτό είναι το καλό νέο. Βέβαια, επιφέρει και σημαντικές διευκρινήσεις στην κατάσταση της Δυτικής Σαχάρας, που εμείς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και τα άλλα θεσμικά όργανα οφείλουμε ομοίω να λάβουμε υπόψη. Και το περιεχόμενο αυτό δηλαδή της ε, αποφάσεως του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Εμπορεύματα που προέρχονταν από τη ε, Δυτική Σαχάρα στο παρελθόν de facto καλύπτονταν από τη συμφωνία. Όμω λέει τώρα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στην απόφαση του Δεκεμβρίου ότι αυτό δεν είναι δυνατόν. Επιβεβαίωσε το Δικαστήριο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να συνάψει συμφωνία με το Μαρόκο που να καλύπτει τη Δυτική Σαχάρα, αλλά αυτό πρέπει να γίνει ρητό και να λάβει υπόψη ορισμένα στοιχεία όπως τη βιωσιμότητα καθώς και ευεργετήματα για τον τοπικό πληθυσμό. Και όπως είπε ο Βίνσεντ έχουν αρχίσει οι διαπραγματεύσεις στο τεχνικό επίπεδο με το Μαρόκο για να καταλήξουμε σε μια κοινή πορεία προς τα εμπρός. Για μας βεβαίως είναι απολύτως ουσιώδες να μην διακόψουμε το, τις εμπορικές ροές με ένα τόσο σημαντικό εμπορικό εταίρο όσο το Μαρόκο. Βεβαίως από την άλλη μεριά είναι αληθές ότι μέχρι τώρα δεν υπάρχει απαγόρευση για εισαγωγέ προϊόντων από την Δυτική Σαχάρα. Το αποτέλεσμα τη αποφάσεως του δικαστηρίου είναι ότι μπορούν μεν να εισάγονται ακόμη τα προϊόντα από την ε, Δυτική Σαχάρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μπορούν όμω να χαίρουν τη προτιμησιακή ε, Θέλω επίση να τονίσω ότι το θέμα αυτό είναι σημαντικό όχι μόνο για το εμπόριο, αλλά έχει επιπτώσει και στην ευρύτερη διμερή σχέση Ευρωπαϊκής Ενώσεως Μαρόκου και πάλι χωρίς λύση στο παρόν πρόβλημα δεν είναι πιθανόν να μπορέσουν να επαναληφθούν σύντομα οι διαπραγματεύσεις για την συμφωνία DCFTA σε βάθος συνολική συμφωνία εμπορικών συναλλαγών. Εγώ δεν είδα καμιά λύση να προτείνετε για την ώρα, ίσως κάτι να μην πρόσεξα από αυτά που είπατε, αλλά βεβαίως θα διεξαχθεί συζήτηση και μετά μπορείτε να επανέλθετε. Τώρα, ο Γενικό διευθυντή Διευθυντής της ε, Ταξούτ, κ. Καστηριανάκη. Ο Βίνσεντ Πικέ αλλά και ο προλαλή σα, ε, τόνισαν την δέσμευση της Υπηρεσίας Εξωτερικών Δράσεων αλλά και τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την συμμόρφωση με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Από τελωνιακή σκοπιά έχουμε μπροστά μας μια απόφαση η οποία διευκρινίζει ότι υπό το ισχύον νομικό πλαίσιο οι τελωνικές αρχές των χωρών μελών οφείλουν να βεβαιώνουν να βεβαιώνονται ότι δεν χορηγείται προτιμησιακή μεταχείριση σε προϊόντα τη Δυτική Σαχάρα όταν εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ορισμένοι μπορεί να θεωρήσουν ότι η απόφαση του δικαστηρίου σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να έρχεται σε εμπορικέ σχέσει με τη Δυτική Σαχάρα. Α μην υπάρξει σύγχυση και επαναλαμβάνω αυτό που είπατε πριν. Αυτό δεν συμβαίνει. Οι εισαγωγέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την Δυτική Σαχάρα είναι απολύτω νόμιμε. Δεν υπάρχει κανένα είδου απαγόρευση. Το μόνο που είπε στην απόφασή του το δικαστήριο είναι ότι δεν υπάρχει νομική βάση για την πρακτική των προηγούμενων ετών με την οποία οι εισαγωγέ από το τμήμα τη Δυτική Σαχάρα που βρίσκεται de facto υπό δικαιοδοσία Μαρόκου αντιμετωπίζονταν ω εισαγωγέ που ε, διέπονται από την Συμφωνία Συνδέσεως Ευρωπαϊκής Ένωση Μαρόκου. Αυτό σημαίνει ότι από τώρα τα τελωνία στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εντοπίζουν εισαγωγέ που ξεκινούν από την Δυτική Σαχάρα, για τα οποία ενδεχομένως, τις οποίες εισαγωγές ενδεχομένως ζητείται προτιμησιακή μεταχείριση παρανόμω από Ευρωπαίου εισαγωγή. Τα συζητήσαμε τα θέματα αυτά με τις τελωνικές υπηρεσίες των χωρών μελών και του ζητήσαμε να κάνουν τι απαραίτητες ενέργειες όπου έχουν εύλογη αμφιβολία σχετικά με την ομιμότητα του ισχυρισμού προτιμιακής μεταχείρισης να χρησιμοποιούν, να προσφεύγουν στις ε, διατάξεις της συμφωνίας για να συνεργάζονται με τους ομολόγους τους στο Μαρόκο και να ζητούν επαλήθευση και πληροφορίες αναφορικά με την προέλευση των εμπορευμάτων. Κάτι που θα επιτρέψει να εντοπίζονται οι σχετικές αποστολές χωρίς να, αναταραχθούν, χωρίς να διαταραχθούν οι νόμιμες ροές. Ελπίζομαι ότι οι εισαγωγεί θα απόσχουν από το να ζητούν προτιμησιακή μεταχείριση. Αντιλαμβανόμεθα ότι είναι γνωστή η ίδια απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στις ενώσεις εισαγωγέων και εξαγωγέων και θα συνεχιστούν οι προσπάθειες μαζί με τις ελληνικές αρχές για να αποφεύγονται οι συγχύσεις και να επιτευχθεί μια ομο, ομοιογενής μια ενιαία στάση απέναντι στις αγωγές από το Μαρόκο. Οι συνάδελφοί μου τόνισαν επίσης ότι κατά την εφαρμογή της αποφάσεως του δικαστηρίου πρέπει να διατηρήσουμε, να διαφυλάξουμε τα εμπορικά και οικονομικά συμφέροντα για την θέση μας στην περιοχή αυτή του κόσμου. Μόλις τόνισα ότι η συνεργασία με τις μαροκινές αρχές είναι σημαντική ώστε να μπορούν τα ευρωπαϊκά τελωνία να εφαρμόζουν τις επόμενες εβδομάδες και μήνες τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και ταυτόχρονα να αποφύγουν οποιαδήποτε περιττή διαταραχή των εμπορικών σχέσεων με το Μαρόκο. Επίσης είναι σαφές ότι συζητήσεις και συνεργασία μεταξύ Μαρόκου και Ευρωπαϊκής Ένωσης... θα είναι απαραίτητες αν θέλουμε να αναζητήσουμε λύση για μακροπρόθεσμο διάστημα. Λύση η οποία θα επιτρέψει τη θέσπιση νομικής βάσεως που να επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, να χορηγεί το πλεονέκτημα της προσημεροτιμησιακής μεταχείρισης για προϊόντα Δυτικής Σαχάρας προς όφελος του τοπικού εκεί πληθυσμού. Όπως είπε ο Βίνσεντ, μαζί με την Υπηρεσία Εξωτερικών Δράσεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διερευνά την δυνατότητα τέτοιας επέκτασης του πεδίου εφαρμογή, ώστε να αναλυθεί κατάλληλη πρωτοβουλία στο εγγύς μέλλον για να δημιουργηθεί η κατάλληλη νομική βάση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλώς, ευχαριστώ πολύ. Ερχόμαστε τώρα στου ευρωβουλευτέ. Έχω 14 ήδη, 15 στον κατάλογο μιλητών, 15, 16, 17. Άλλος, ποιος προτείνει παραπάνω. Λοιπόν, προτείνω δύο λεπτό καθένας για να μπορέσουμε να τους ακούσουμε όλους. Αρχίζουμε λοιπόν με τον Αντιπρόεδρο της Αντιπροσωπείας για τις σχέσεις μας με τις χώρες Μαγκρέπ. Χιμένες, παρακαλώ, κύριε Χιμένες Παρπά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Οι σχέσεις μας με το Μαρόκο είναι ζωτικές σημασίας για την Ευρώπη Πρώτα απ' όλα, και επειδή εγώ είμαι Ισπανίδα, δίπλα στο Μαρόκο, δηλαδή είναι η χώρα μου, για μένα έχουν μεγάλη σημασία. Είναι πολύ σημαντικό επίσης να σημειώσουμε και ότι έγινε πρόοδος τα τελευταία χρόνια, κάτι το οποίο έχουν χαιρετήσει όλες οι χώρες μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο λοιπόν αποφάσισε, όπως ακούσαμε το Δεκέμβριο, ότι η Αγροτική Συμφωνία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Μαρόκο ισχύει δεν μπορεί να εφαρμοστεί στη Δυτική Σαχάρα. Αλλά ισχύει. Και δεν μπορεί να εφαρμοστεί εκεί εξαιτία τη σύγκρουση που δεν λέει να πάψει. Πρέπει λοιπόν την απόφαση του δικαστηρίου να τη σεβαστούμε, γιατί όπως λένε και οι άλλες χώρες στο Μαγκρέμπ, είναι πολύ σημαντικό να τηρηθεί η απόφαση αυτή για όλους. Τώρα συγχρόνως έχουμε και εταιρική σχέση και όπω λέει η απόφαση αυτή ισχύει. Πράγμα που σημαίνει ότι μπορούμε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε βάσει τη συμφωνία αυτή, στηρώντα βέβαια πάντα τη διεθνή νομιμότητα. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να χρησιμοποιήσει ό,τι μηχανισμού μπορεί έτσι ώστε να επιτευχθεί πρόοδο και ευημερία στην περιοχή αυτή του Μαγκρέμπ που έχει μεγάλη σημασία για του Ισπανού και του Ευρωπαίου. Η Δυτική Σαχάρα και το Μαρόκο πρέπει να βρουν ένα πλαίσιο πέρα από ό,τι παλιό γνωρίζαμε που θα τους επιτρέψει να κινηθούν μαζί και να πετύχουμε τέλος κάτι στην Ευρώπη μετά από τόσες συγκρούσεις. Πρέπει να καταλήξουμε σε μία κατάσταση από την οποία όλοι να έχουν να κερδίσουν. Win-win όπω είναι τη μόδα να λέμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιλαμβάνεται το σημαντικό ρόλο που παίζει το βασίλειο του Μαρόκου στην περιοχή και γι' αυτό και θα το στηρίξει το Μαρόκο προκειμένου να καταλήξει να βρει λύσει για τον πληθυσμό τη Δυτικής Σαχάρα, μια λύση με την οποία να συμφωνούν βέβαια και εκείνοι και έτσι να μπορεί να γίνει εκμετάλλευση των πόρων του. Πολιτική συμφωνία δίχω άλλο και η Ευρωπαϊκή Ένωση ελπίζω να μπορέσει έτσι να εξομαλύνει τις σχέσεις της με την περιοχή αυτή που όσο περνά ο καιρός όλο και πιο κοντά στην Ευρώπη βρίσκεται. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα πάμε στην ομάδα του ΕΛΚ. Ο κύριος Μιλανμόν έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πολύ στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης αλλά και τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρώτα απ' όλα θέλω να επαναλάβω αυτό το οποίο έχω πει και σε άλλη συζήτηση που κάναμε εδώ τον Ιανουάριο για την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου του Δεκεμβρίου που διατηρεί την ισχύ της συμφωνίας αυτής με το Μαρόκο και ακυρώνει την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου του 2015. Το Συμβούλιο είχε προσφύγει κατά της πρώτης απόφασης αυτής του Γενικού Δικαστηρίου. Επιτρέψτε μου λοιπόν, Πρόεδρε, εδώ να σας μεταφέρω κάποιες σκέψεις. Πρώτα απ' όλα, η σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Μαρόκο είναι θεμελιώδου σημασία και πρέπει να την φροντίζουμε γιατί είναι τέρος προνομιακός μάλιστα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ιδιαίτερα προχωρημένο καθεστώς όσον αφορά τι σχέσει μας. Δεύτερον, η Δυτική Σαχάρα μπορεί να βρει λύση μέσα από τον ΟΗΕ και μέσα από τις διμερείς ε, σχέσεις ανάμεσα στο Μαρόκο και το Πολυσάρι υπό την αιγίδα βέβαια του ΟΗΕ. Εμείς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να προσπαθήσουμε το ζήτημα της Δυτικής Σαχάρας που αλλού λύνεται να μην παρεμβαίνει στις διμερείς σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Μαρόκο. Πολύ σημαντικές σχέσεις, είπαμε, είναι προνομιακός εταίρος το Μαρόκο για μας και συμφωνούμε όλοι σε αυτό. Είναι μια σχέση όχι μόνο ε, εμπορική ή ε, πολιτική αλλά και ασφάλειας για να καταπολεμήσει στην τρομοκρατία, ε, το μεταναστευτικό κτλ. Εξάλλου το Μαρόκο μετά τόσα έγιναν με την Αραβική Άνοιξη αποτελεί σημείο αναφοράς σταθερότητας και ήσυχης δύναμης που προχωράει προς τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ελευθερίες. Συνεπώ, αυτό που θέλω είναι να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικών δράση, να βρούνε τρόπου για να λυθεί το ζήτημα αυτό, λαμβάνοντα υπόψη και σεβόμενη φυσικά πάντα την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, αλλά να βρεθεί ένας τρόπος ε, με τον οποίο να μην αλλοιωθούν οι σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Μαρόκο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο κ. Παγνιό για τον λόγο. Οι σοσιαλιστές ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τέσσερα σχόλια έχω στα πλαίσια της Καταρχήν, έχουμε απόφαση του ΔΕΚ περίπλοκη. Και στη η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Μαρόκο. Και το βάζει σε ίδιο επίπεδο Πολυσάριο και η Αλγερία. Δεν κέρδισε το Πολυσάριο πολύ, διότι ισχύει η απόφαση του 2012. Η απόφαση είναι σαφέστατη όσον αφορά τη μη εφαρμογή στην επικράτεια τη Δυτική Σαχάρα. Η απάντηση τη Ένωση σε αυτή την κατάσταση που είναι πάρα πολύ περίπλοκη δεν μπορεί να είναι απλουστευτική, όπως είδαμε σε αυτά που ακούσαμε προηγουμένως στην αρχή της συναντήσεως. Μετά, δεύτερο σχόλιο, τα διεθνή κείμενα μπορεί να διατηρηθούν σε σχέση με το Μαρόκο, διαβάζοντας υπόψη την απόφαση του ΔΕΚ. Όπως το πρωτόκαλο Αλίας που υιοθετήθηκε το 2013 προβλέπει τη συμπερίληψη της Σαχάρας στη Συμφωνία και προβλέπει νομικές διατάξεις για τις ντόπιου που ευνοούν τους ντόπιου πληθυσμού. Και έχουμε ήδη εμπειρία της εφαρμογής της α, αποφάσεως. Μπορούμε να ξεφύγουμε τα διέξοδο χωρίς να βλάψουμε τις σχέσεις με το Μαρόκο. Τρίτον, εκείνοι που θέλουν να μεταρρυθμίσουν το κοινοβούλιο μας σε συνέλευση του Συμβουλίου Ασφαλείας στο ΙΕ πρέπει να προσέξουν. Μόνο στον ΙΕ θα βρεθεί μια βιώσιμη και δίκαιη λύση αποδεκτή από όλους δεν ωφελούνται οι τόποι πληθυσμοί και η τοπική σταθερότητα διαφορετικά. Θα πρέπει να αποφύγουμε πολιτική τοποθέτηση. Στην Τάλα είχα συμμετάσχει στη διάσκεψη και συζητήσεις είδαμε ότι εξελίσσεται μετά από ότι ήταν έρημο Σαχάρα, εξελίσσεται οικονομικά και κοινωνικά προς όφελος των πληθυσμών. Θα πρέπει να τη διαφυλάξουμε την περιοχή, δίνοντας ένα καθεστώς. Πραγματικό ερώτημα. Πώς μπορούμε να δράσουμε. Πώς μπορούμε να χρησιμεύσουμε στον ΟΗΕ και το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Θα πρέπει τις επόμενες εβδομάδες να διευκολύνουμε τις διαπραγματεύσεις και τις συζητήσεις. Ευχαριστώ. Ο κ. Βίστεζεν, αντιπρόεδρος της Επιτροπής μας, εκπρόσωπος του ECR. Ήδη υπογραμμίστηκε από αρκετού συναδέλφου. Ο κ. Βίστησεν είναι σημαντικότατο σύμμαχο για την Ευρώπη, το Μαρόκο. Σημαντική χώρα για τη γειτονιά, για το εμπόριο, για την ασφάλεια, για την καταπολέμηση της νομοκρατίας. Συνεπώς είναι πολύ σημαντικό να επιληθεί το θέμα της αποφάσεως του 10. Από τη μια πλευρά αναφυσβήτητα πρέπει να λάβουμε στα σοβαρά υπόψη αυτή την απόφαση και να την αντιμετωπίσουμε και να εφαρμόσουμε συγκεκριμένα. από την άλλη, χαίρομαι που ακούω που τα μέλη τη Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζουν πραγματιστικέ ε, λύσει. Φερρυπίν, κατονομάζοντας τη Δυτική Σαχαρά, θεωρώντα σαν επικράτεια και προσπαθούν να βρουν μια συμφωνία με τις αρχές του Μαρόκου. Δεν ωφελείται η ειρηνευτική λύση εάν επιβάλλουμε πιο αυξημένου δασμού στη Δυτική Σαχάρα από ό,τι στο υπόλοιπο Μαρόκο, από ό,τι στο Μαρόκο. Και να αφήσουμε να ανθίσει περισσότερο το υπόλοιπο Μαρόκο και η Δυτική Σαχάρα. Είναι πολύ ευαίσθητο πρόβλημα. Η λύση πρέπει να βρεθεί στον ΟΗΕ. Όχι σε διμερείς σχέσει μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Μαρόκου. και υποστηρίζω τις προσπάθειες της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρέπει να συμμορφωθούν οι φορείς με την απόφαση του ΔΕΚ και απ' την άλλη να προχωρήσουμε με πραγματιστικό τρόπο. Με τρόπο εποφελή για τις διμερείς μας ε, σχέσεις και για τους ε, λαούς της ε, Δικής Σαχάρας. Για τους πράσινους, ο κ. Μπούχνερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Τρεις ερωτήσεις. Ευχαριστώ και τρεις ερωτήσεις. Πρώτα, είπατε ότι διαπραγματεύεστε με τους ανθρώπους του Πολυσάριο. Εγώ θυμούμαι ότι αυτή είναι η μόνη αναγνωρισμένη εταίρη για τις διαπραγματεύσεις αυτές. Σας το υπενθυμίζω μάλλον αυτό. Να μου πείτε κάτι παραπάνω. Δεύτερη ερώτηση. Μιλούμε πολύ για την συμπερίληψη της Δυτικής Σαχάρας στις συμφωνίες μας κλπ. Τι σημαίνει όμως Δυτική Σαχάρα. Σημαίνει τους ανθρώπους που διαβιούν εκεί, σημαίνει τους επίκους, επίκους από το Μαρόκο ή, ή τους γνήσιους Δυτικοσαχαριανούς. Νομίζω ότι υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη διάκριση, διότι τις παρατηρήσεις που άκουσα προηγουμένως Ελέγχθη δηλαδή ότι χρειάζεται να συνεχίσουμε. Υπάρχουν όμως μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν κατασταθεί τώρα από το Μαρόκο, που έχουν εγκατασταθεί σε εδάφη της Δικής Σαχάρας. Πρέπει να κάνουμε τη διάκριση εκεί και να δώσουμε την προτίμηση στους γνήσιους δυτικοσαχαριανούς κατοίκους. Δεύτερο, εισαγωγές τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση εισάγουμε μόνο από συγκεκριμένε χώρε. Η Δυτική Σάχαρα δεν περιλαμβάνεται σε αυτέ. Οι εισαγωγέ από την, περιφερεια, την περιοχή αυτή είναι κατά τη γνώμη μου παράνομε. Δεν ήθελα πολύ να σχολιάσετε και αυτό. Σας ευχαριστώ. Ξέχασα μία ομάδα, ζητώ συγγνώμη. Η κυρία Ντεζανέ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους όσους πήραν το λόγο. Να πω δύο-τρία πράγματα, απλούστατα. Καταρχά, πιστεύω ότι είναι μεγάλο το διακύβευμα. Πρέπει να έχουμε καλέ σχέσει μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Μαρόκου. Και αυτέ οι καλέ σχέσει, κατά την άποψή είναι πρώτα απ' όλα πολιτικέ πριν από εμπορικέ. Έχουμε κοινά συμφέροντα. Έχουμε κοινά συμφέροντα όσον αφορά την ειρήνη, την ασφάλεια, την καταπολέμηση τη τρομοκρατία. Έχουμε κοινά συμφέροντα στον τομέα τη μεταναστεύσεω και θα πρέπει να διατηρήσουμε σε θυσία αυτή τη ε, σχέση. Το δεύτερο, εμπορικές σχέσεις. Προφανώς, όπως είπε ο Ζιλπανιό, δεν είμαστε όλοι εδώ. Δεν θα ρυθμίσουμε εδώ το θέμα της Δυτικής Σαχάρας. Χρειάζεται μια προσέγγιση πιο συγκεκριμένη που διευκολύνει την κατάσταση. Άκουσα κάποια τροπολογία για την κάποια αλλαγή της γεωργική Συμφωνίας. Δεν ήθελα να ξέρω περισσότερα γι' αυτό. Και σαν εισηγήτρια για τις γεωγραφικέ ενδείξεις, στα πλαίσια της γεωργία ψηφίσαμε στην Επιτροπή Ίντα μια έκθεση μέσα Ιουνίου. Έχουμε. Θα ψηφίσουμε για τι ε, ενδείξει γεωγραφική προελεύσης όσον αφορά ε, τι εμπορικέ σχέσει Ευρωπαϊκή Ενώσης ω Μαρόκου. Πρέπει να ξέρω πού βρισκόμαστε. Είπατε ότι θέλουμε συγκεκριμένε λύσει. Κάποιοι είπατε δεδειγμένε λύσει, αλλαγέ. Ποιο είναι το πρόγραμμα, κατά την άποψή σα, για τι συγκεκριμένε λύσει. Συμφωνούν τα διάφορα κόμματα με αυτέ τι λύσει. Προφανώ η Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, επίση το προτείνουμε, είναι ανοιχτό ο διάλογο πάνω σε αυτέ τι ρεαλιστικέ λύσει με το Μαρόκο. Αυτή είναι η ερώτηση. Ευχαριστώ. Η κυρία Μπεγκίν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συνάδελφοι, ε, μέσα στο κίνημα των πέντε αστέρων πάντα ήμασταν αρκετά επικριτικοί όσον αφορά τη συμφωνία με το Μαρόκο. Λόγω των σοβαρών συνεπειών που έχει για τι μεσογειακές χώρε, οι γεωργοί, μα ξέρουν τι πράγμα αναφέρω. Ένα παράδειγμα. Από το Δεκέμβριο 2015 με Ιανουάριο του 2016, τα, οι ντομάτε αυξήθηκαν κατά 74%. Ε, εισαγόμενα στην Ιταλία και κατέρευσε η Ιταλική αγορά σοφορά αφορά τα προϊόντα αυτά. Και το ίδιο και για τα πορτοκάλια. Ε, ζητήσαμε λοιπόν να εφαρμοστεί ρήτα διαφύλαξη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν θα έπρεπε να μπουν αυτά τα προϊόντα. Γονάτισε αυτό το μέτρο του γεωργού μα και δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Λοιπόν, το ΔΕΚ αποφάσισε ότι η συμφωνία δεν ισχύει για την επικράτεια της Δυτικής Σαχάρα. Δεν θέλω να επισέλθω τώρα σε νομικές λεπτομέρειες αποφάσεω ή την έφεση. Αλλά επιβάλλονται κάποια καθήκοντα από αυτή την απόφαση. Αν δεν ισχύει η συμφωνία πρώτα απ' όλα, θα πρέπει να εντοπιστούν ποια εμπορεύματα και ποια εμπορεύματα ε, προέρχονται από τι αποκλεισμένε περιοχέ και να αποκλειστεί η εισαγωγή του. Τα στοιχεία δεν είναι ακριβή όμω Η παραγωγή στη Δυτική Σαχάρα το ντομάτα είναι από 0,01% μέχρι 70% της παραγωγής συνολικής του Μαρόκου. Χωρίς να μετρήσουμε ότι το Μαρόκο σχεδιάζει μέχρι το 2020 να αυξήσει σε αυτές τις περιοχές άλλες ε, πάρα πολλά απορκευτικά. Λοιπόν, έχουμε και ψάρια που εξάγονται κλπ. Και, και θα πρέπει όλα τα προϊόντα να εξεταστούν. Λοιπόν, πώς προτίθεται να εξετάσει αυτό το θέμα, θα εφαρμόσει πιο καθεστώς τους κανόνες ε, προέλευσης των προϊόντων. Ε, άλλο μέτρο, θα υπάρχει άλλη τικετοθεσία χρησιμοποιώντας διαφορετικούς τελωνιακούς κώδικες για τα προϊόντα από την περιοχή αυτή. Ε, κάτι πιο πρακτικό. Αν η Γεωργία και λύση της Ευρώπης έχουν ζημιωθεί λόγω μιας συμφωνίας που αποκαλύφθη ότι εν μέρη είναι παράνομη θα πρέπει να εκτιμήσουμε ποια είναι αυτή η ζημιά και ενδεχομένω δοθούν αποζημιώσει. Λοιπόν, θα ήθελα να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν αξιολόγησε αυτή την επιλογή, εάν θα δώσει κάποιε αποζημιώσει και αν δώσει αποζημιώσει και χρήματα, μέχρι πότε θα τα δώσει. Ευχαριστώ. Ο κύριο Μπουργκέζιο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, πάρα πολύ γρήγορα. Σίγουρα, στη βάση υπάρχει κάποια επίκριση. Κυρίως από πλευρά εμάς που εκπροσωπούμε τους Ευρωπαίους παραγωγούς. Διότι έχουμε να κάνουμε με μια συμφωνία που περιέχει πτυχές πολύ περίπλοκες και σκοτεινές. Χρειάζεται να ρίξουμε φως. Τα νομικά προβλήματα που απορρέουν από την απόφαση του ΔΕΚ πρέπει να κατανοήσουμε καλύτερα αν αυτή η απόφαση εμποδίζει τις αγωγές προϊόντων με προέλευση τη Δυτική Σαχάρα. Διότι αυτό δεν μου φαίνεται πάρα πολύ σαφές. Γιατί αυτή η περιπτώση θα ήθελα να γνωρίζω ποια είναι η ακριβής θέση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και ποιε πρωτοβουλίες νομικής φύσεως ε, έχουν δοθεί, ποιε νομοδοτήσει νομικέ έχουν δοθεί. Είναι πολύ σημαντικό για να αξιολογήσουμε πληρέστερα τη συμφωνία με το Μαρόκο. Επογραμμίσουμε ότι το νομικό καθεστώς της Δυτικής Σαχάρας δεν θα πρέπει να βλάψει τη σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης Μαρόκου. Είναι ξεχωριστό θέμα, εκτός των αρμοδιοτήτων μας. Είναι θέμα που αφορά αποκλειστικά την αξιολόγηση και την παρέμβαση των Ηνωμένων Εθνών. Thank you. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Αλαφράγκα τώρα, εκ μέρους του ΕΛΚΑ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Οι συνεδρίες αυτές της ε, ΑΦΕΤ είναι αναγκαίες και καλώς γίνονται με τους εταίρους μας μας ε, υπενθυμήθηκε ποια είναι η απόφαση αυτή του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που έχει επιπτώσεις και βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Είπανε και άλλοι πώς θα διατηρήσουμε τις σχέσεις μας με τον εταίρο μας αυτό που είναι το βασίλειο του Μαρόκου που είναι προνομιακός εταίρος και πώς θα εφαρμοστεί η απόφαση αυτή. Ακούσαμε διάφορα αλλά αυτό που θα ήθελα να ξέρω, πριν φύγω την πράγμα και σε άλλη είναι τι γίνεται με τη συμφωνία σύνδεση. Πρέπει να αλλάξει η εμπορική συμφωνία, η γεωργική για την προέλευση. Χρειαζόμαστε νέε κατευθυντήριε γραμμέ για την πραγμάτευση. Και πώ θα συμφιλιώσουμε όλη αυτή τη διαδικασία που κρατάει χρόνο, χωρί να διακινδυνεύσει η ροή εμπορικών προϊόντων με το Μαρόκο, που μειώθηκε πάρα πολύ το τελευταίο χρόνο και δεν μπορούμε να το αφήσουμε να συνεχίζεται αυτό. Και πώς θα εφαρμοστεί η απόφαση αυτή λοιπόν στα εδάφη της Δυτικής Σαχάρας. Αν λοιπόν στη Δυτική Σαχάρα εφαρμόσουμε προτιμησιακή μεταχείριση, αυτό συνάδει με την προτιμησιακή μεταχείριση που προβλέπει η συμφωνία μας με το Μαρόκο ή πρέπει να υπάρξει ειδικό καθεστώς όπως προβλέπεται για τη Μολδαβία και την Ουκρανία Επιμένω ότι το σημαντικό είναι να μην πληγεί η ροή εμπορικών προϊόντων μεταξύ Μον και του Μαρόκο και χωρίς φυσικά να πληγεί ο κόσμος που βρίσκεται στη Δυτική Σαχάρα. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Οι σοσιαλιστές. Η κυρία Βίνα τώρα. Η κυρία Ρένα. Ευχαριστώ. Θα επαναλάβω δύο αρχές. Ότι η συζήτησή μα πρώτα απ' όλα δεν αμφισβητεί τη σημασία που έχουν διπλωματικέ πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές σχέσεις ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Μαρόκο. Και δεύτερον, δεν σκοπεύουμε εδώ να λύσουμε την ε, σύγκρουση όσον αφορά τη Δυτική Σαχάρα. Υπάρχει άλλο βήμα γι' αυτό που είναι τα Ηνωμένα Έθνη. Ρόλος μας, μόνο που είμαστε Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι να εφαρμόσουμε τις εμπορικές μας συμφωνίες με το Μαρόκο βάσει της συμφωνίες του δικαστηρίου. Πρώτα απ' όλα της απόρριψης της ανέρεσης και δεύτερον να μην εφαρμόζεται η συμφωνία αυτή στη Δυτική Σαχάρα. Συνεπώς, αποκλείει τη Δυτική Σαχάρα το δικαστήριο και αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούν να υποφεληθούν προϊόντα από τη Δυτική Σαχάρα με προτιμησιακούς ε, τελωνιακούς δεσμούς. Λοιπόν, πρώτον, πώς θα εντοπιστούν τα προϊόντα αυτά, πώς θα γίνουν η έλεγχη, αν όντως αυτό ακολουθήσουμε. Αλλά από ό,τι κατάλαβα, εσεί προτείνετε κάτι άλλο. Προτείνετε να τα συμπεριλάβουμε τα προϊόντα από τη Δυτική Σαχάρα. Υποθέτω ότι αυτό το στηρίζει και το Μαρόκο. Αυτό σημαίνει όμως ότι πρέπει να τροποποιηθεί η συμφωνία και ακούσαμε ότι η Επιτροπή θέλει μια τροπολογία. Ζητάει όμως επίσης να υπάρξει και μια αρχή συνένεσης και επιστροφής στον πληθυσμό. Δηλαδή απέναντι στο Πολυσάριο ρωτάω γίνεται συζήτηση για τη συνένεση αυτή που πρέπει να δοθεί και για την επιστροφή των κερδών, υποθέτω, στον πληθυσμό. Υπάρχει επίσης και η λογική αποκλεισμού των προϊόντων από τη Δυτική Σαχάρα, κάτι το οποίο ισχύει από πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών στην δικιά του συμφωνία με το Μαρόκο. Πώς εφαρμόζουν αυτόν τον αποκλεισμό των προϊόντων από τη Δυτική Σαχάρα οι Ηνωμένε Πολιτείε, πολύ θα ήθελα να το ξέρω. Και τέλος πρέπει να δουλέψουμε και προληπτικά όσον αφορά τις συμφωνίες ε, σύνδεσης για να δούμε πώς και πότε θα μπορέσουμε και εμείς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αποφασίσουμε. Πρόεδρο ευχαριστούμε. Η κυρία Φωτίνκα τώρα, εκ μέρους του ΙΣΙΑΡ, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ όλους ε, τους προσκεκλημένους μας που πήραν το λόγο. Θέλω να υπογραμμίσω ότι το Μαρόκο δεν είναι μόνο ε, από τους πιο μεγάλους μας εταίρους όσον αφορά το εμπόριο αλλά και την ασφάλεια, συγχρόνως παίζει έναν ε, πολύ σημαντικό σταθεροποιητικό ρόλο στην περιοχή. Και όχι μόνο γιατί ελέγχει τις μεταναστευτικές ροές, αλλά γιατί επίσης αντιμετωπίζει και τις βαθύτερες αιτίε της μετανάστευσης. Άρα ο ρόλος του βασιλείου του Μαρόκο στην περιοχή είναι πάρα πολύ σημαντικός και πολύ θετικός. Πρέπει να παραδεχτώ ότι έχω κάποιες ανησυχίες για την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Γιατί για μένα έμεσα ανακατεύεται στο θέμα της δικαιοδοσίας του Μαρόκο στα εδάφη της Δυτικής Σαχάρας. Πράγμα το οποίο κανονικά είναι αρμοδιότητα των Ηνωμένων Εθνών. Οπότε να ρωτιέμαι, είναι δυνατόν να έχουμε το κείμενο της απόφασης με την αιτιολόγηση αλλά και την γνωμοδότηση του Γενικού Εισαγγελέα για το θέμα αυτό. Ευχαριστούμε κυρία Φωτίγκα. Η απόφαση από ό,τι μου να είναι, έχει δημοσιοποιηθεί online, μπορείτε να τη βρείτε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Τώρα, η κυρία Βαλέρο. Ευχαριστώ. Συμφωνώ με αυτά που υπόθηκαν. Παρακαλώ βάζετε τα ακουστικά σας. Λοιπόν, άκουσα αυτά που υπόθηκαν και παρατηρώ ότι όλοι λησμόνησαν ότι εδώ μιλάμε για 40 χρόνια που υπάρχει αυτό το πρόβλημα κατοχής της Δυτικής Σαχάρας του πλευράς του Μαρόκου. Εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση παίρνουμε τελικά τη θέση του κατακτητού και όχι τη θέση του κατακτημένου. Και αυτό είναι πραγματικά αρνητικό. Διαβάζοντας τη μελέτη που εξεπονήθη, Σημειώνω ότι ξεκινά από την υπόθεση ότι δεν, μπορεί να υποστη... δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε εκείνον που κατέχει το έδαφος. Μπορούμε να συνεργαζόμαστε με το Μαρόκο χωρίς να μιλάμε για τα προϊόντα που προέρχονται από τη Δυτική Σαχάρα. Είναι παράλογο να υποστηρίζουμε εκείνον που είναι ο κατακτητής και όχι τον κατακτημένο δεν θα αγοράζαμε ποτέ τα προϊόντα της Δυτικής Σαχάρας αν τηρούσαμε το ε, διεθνές δίκαιο. Θα πρέπει να λυθούν όλα αυτά. Ο πληθυσμός της Δυτικής Σαχάρας πρέπει να μπορεί να, έχει, να, να εκμεταλλεύεται το εμπόριο των δικών του προϊόντων και δεν θα πρέπει να αποφελούνται οι έπικοι της περιοχής που έρχονται από το Μαρόκο στη Δυτική Σαχάρα. Έχουμε το, φρόντε, το μέτωπο Πολυσάριο που εκπροσωπεί τη Δυτική Σαχάρα. Θα πρέπει να αποφασίσουμε αν θέλουμε να συνεχίσουμε το εμπόριο με την περιοχή της Δυτικής Σαχάρας. Θα θέλουμε μια συμφωνία, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαπραγματευτεί αυτή την περιπτώση με το μέτωπο Πολυσάριο. Όλα τα κράτη-μέλη υποστηρίζουν την ιδέα ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί η απόφαση. Αλλά αυτό είναι παράλογο. Πρέπει να δημιουργήσουμε δηλαδή δημιουργικές λύσεις. Αναφέρεται η Δυτική Σαχάρα. Το μέτωπο Πολυσάριο θα πρέπει να, θα πρέπει να αποτελέσει ένα συνομιλητή μας. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Καστάλντο από το EFTD τώρα παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ εκπλήσωμαι κάπως, διότι ακούγοντας τη συζήτηση τη σημερινή έχω την εντύπωση ότι εδώ ε, λέμε ότι η πραγματικότητα πρέπει να προσαρμοστεί στη συμφωνία μας και όχι η συμφωνία μας να προσαρμοστεί στην πραγματικότητα. Και τη νομική πραγματικότητα και την de facto πραγματικότητα. Λέει η απόφαση του ΔΕΚ σαφώ ότι η Δυτική Σαχάρα δεν ανήκει στο βασίλειο του Μαρόκου, σύμφωνα με το διεθνέ δίκαιο. Αυτή δεν είναι μια πολιτική μάχη, είναι ένα θέμα νομικό. Κανένα δεν θέλει να αμφισβητήσει τη σημασία των σχέσεων με το Μαρόκο, Μαρόκο από όλε τι πλευρέ. Θα πρέπει όμω να λάβουμε υπόψη ότι είμαστε ένα κράτο δικαίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κράτο δικαίου ε, και θα πρέπει να σέβεται τι αποφάσει. Πάνω σε αυτό λοιπόν έχω δύο ερωτήσει. κετοθεσία. Από πλευρά τη αποφάση του 106 υπογραμμίζεται σαφώ ότι οδήποτε εμπόριο γεωργικών αγαθών χωρί τη συνένεση των Σαχράουι είναι παράνομο. Δεν έχει νομική δυνατότητα να βάλει πιστοποιητικά σε αυτά τα προϊόντα που παράγουν στη Δυτική Σαχάρα, το Μαρόκο. Εάν βάλουμε την κοιτοθεσία όπως προτάθηκε πριν, όχι μόνο είμαστε κάπως παράνομοι, αλλά πάνω απ' όλα δεν λύνεται το πρόβλημα τελικά του δικαιούχου. Διότι πολλοί μιλήσαν για την ανάπτυξη την οικονομική της περιοχή. Το θέμα είναι ότι αυτή η ανάπτυξη δεν ωφελεί τους πολίτες τη περιοχή σύμφωνα το διεθνές δίκαιο. Και ένα μεγάλο ποσοστό αυτών είναι πρόσφυγες εδώ και πολλές δεκαετίες. Δεύτερο σημείο και πάω στο άλλο ερώτημα εξ αυτού. Το θέμα της συνενέσεως του μετόπου Πολυσάριο. Σύμφωνα το σημείο 105 τη απόφασης που αναφέρεται στην, στην 34-37 απόφαση του ΟΗΕ, το μέτωπο Πολυσάριο εκπροσωπεί τη Δυτική Σαχάρα. Συνεπώ, η μοναδική λύση εφικτή για να διευρυνθεί αυτή η λύση είναι να συμπεριληφθεί και το μέτωπο Πολυσάριο, να βρεθεί μια λύση που πραγματικά να είναι υποφελή για τον πληθυσμό τη Σαχάρα. Κλείνω ότι θα πρέπει να δοθεί μια απάντηση, όπω είπε άνθρωπος Μπεγκέν, για του αλληλεί και του γεωργούς του Ευρωπαίου και για το μέτωπο Πολυσάριο, για τη ζημιά που έχουν υποστεί οι ντόπιοι παραγωγοί. Οι αποφάσει δεν αλλάζουν, δεν επανερμηνεύονται, δεν επανεφευρίσκονται, ε, τι σέβονται τι αποφάσει και τι εφαρμόζουν τι αποφάσει κανονικά. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε τέσσερις ομιλητές που να Σε υπενθυμίσω ότι θα πρέπει να ολοκληρώσουμε αυτό το σημείο στις 4 και 4. Πριν μιλήσουν οι τέσσερις συνάδελφοι, θα θέλαμε να ακούσουμε και μερικές απαντήσεις τουλάχιστον από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τέσσερις τελευταίοι συνάδελφοι, παρακαλώ να είστε τηλεκονικοί. Η κυρία Ροτρίγκε Πινέιρο είναι η επόμενη. Ευχαριστώ πολύ και τους δύο πρόεδρους μας και ευχαριστώ πολύ και τους εκπροσώπους της υπηρεσίας εξωτερικών σχέσεων, τη Κομισιόν κτλ. Συμφωνώ με τα όσα ακούσαμε για το ότι είναι πολύ σημαντικό να διατηρήσουμε πάρα πολύ καλές σχέσεις ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Βασίλειο του Μαρόκου. Άρα πρέπει να βρεθεί μια νομική λύση η οποία να πάψει να μας έχει στην αβεβαιότητα που μας έχει σήμερα. Πρέπει να βρεθεί μια ισορροπημένη λύση μεταξύ όλων των διαφερόμενων πλευρών που να στηρίζει βέβαια όλους τους εμπλεκόμενους. Να δούμε μετά την απόφαση πώς θα προχωρήσουμε σεβόμενοι πάντα τα δικαιώματα όλων των πλευρών, το διάλογο, την αρχή της διαβούλευσης αλλά και της συνένεσης. Η ερώτησή μου είναι η εξή όσον αφορά τη σημερινή κατάσταση. Είναι ξεκάθαρο ότι η απόφαση αυτή ε, αποκλεί τις εμπορικές σχέσεις ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Δυτική Σαχάρα από τη συμφωνία την εμπορική Ευρωπαϊκής Ένωσης Μαρόκο, γιατί είναι διαφορετικό το τελωνιακό καθεστώς, οπότε εγώ ρωτάω πώς μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι η εξαγωγή αγροτικών προϊόντων. Οποροκυπευτικά που με ενδιαφέρουν εμένα. Πώς μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το ότι τέτοιο προκυπευτικά που παράγονται στη Δυτική Σαχάρα δεν θα φτάνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση με το προνομιακό καθεστώς εφόσον θα μπορούν να περνάνε μέσα από το Μαρόκο. Μπορούμε να το ξέρουμε κατά πόσο τελικά εφαρμόζεται πραγματικά η απόφαση αυτή του δικαστηρίου ή όχι. Και πώς θα ενημερωνόμαστε για όλη τη διαδικασία διαπραγματεύσεων. Θέλω διαφάνεια, ακριβώς γιατί το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Γιούρεκ τώρα, εκ μέρους του ECR, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Η τεράστια πλειοψηφία των συναδέλφων τόνισαν, τόνισε ότι οι σχέσεις με το Μαρόκο είναι σημαντικότατες. Πολύ σημαντικές για την Ευρώπη το Μαρόκο δεν είναι μόνο σημαντικός παράγων σταθερότητος και ασφαλείας στην περιοχή, αλλά πρέπει να θυμόμαστε ότι οι οικονομικές και οι πολιτικές σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης είναι σημαντικότατες για τη σταθερότητα στη χώρα αυτή και δεν θα πρέπει να υπονομεύονται αυτές οι συνθήκες. Βεβαίως η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου θα πρέπει να εκτελεστεί να γίνει σεβαστή, όμως θα πρέπει να εφαρμοστεί με τρόπο τέτοιο που να μην βλαφτούν τα συμφέροντα των εταίρων μας. Πολλοί συνάδελφοι ανέφεραν ότι διαρκεί περίπου 40 χρόνια αυτή η κατάσταση, αυτή η σύγκρουση. Δεν αφορά μόνο το μέτωπο Πολυσάριο και το Βασίλειο του Μαρόκου, Άρα είναι μια διεθνή σύγκρουση που εμπλέκει και πολλές γειτονικέ χώρες. Και γι' αυτό θα πρέπει να σκεφτούμε τα θέματα ασφαλείας, της ασφαλείας της Ευρώπης, της ασφαλείας των φίλων μας. Γνωρίζουμε ότι η ασφάλειά μας κλονίστηκε πολύ από την κατάσταση που επικρατεί στη Λιβύη και θα δεν θα ήταν πολύ συνετό να διαταράξουμε τη σταθερότητα ή ασδήποτε χώρας εταίρου με την οποία να απολαμβάνουμε πολύ καλές σχέσεις. Κάτι που ισχύει με το Μαρόκο. Θα ήταν αντιπαραγωγικό κατά των συμφερόντων μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσεως. Οι εκπρόσωποι της υπηρεσίας αυτής φαίνεται ότι προσπαθούν να βρουν λύση. Θέλουμε να σεβαστούμε το κράτος δικαίου, ταυτόχρονα όμως δεν πρέπει να υπονομεύουμε και τη συνεργασία μας. Αυτό θα πρέπει να το έχουμε υπόψη. Ευχαριστώ. Η κυρία Χάουταλα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σύντομη ερώτηση. Η υπηρεσία εξωτερικής δράσης βλέπει ότι ίσως μπορούμε να είμαστε διαμεσολαβητής η Ευρωπαϊκή Ένωση μεταξύ των εκπροσώπων της ε, Δυτικής Σαχάρας, δηλαδή του μετώπου Πολυσάριου και του Μαρόκου. Η κυρία Βαλέρο αναφέρθηκε σε μια μελέτη. Θεωρούμε ότι δεν είναι καθόλου επαγγελματική αυτή. Πολύ ερασιτεχνική. Ατεκμηρίωτη. Καλύτερο θα ήταν πριν δημοσιευθεί η μελέτη να εξεταστεί από πλευράς νομικής προσεκτικότατα. Καλώς. Θα επανέλθουμε σε αυτό σε λίγο. Ο κύριος Ματσολέζη. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα πρέπει να διαβάσουμε. Να διαβάσουμε την απόφαση του δικαστηρίου που δεν μιλάει για μια κατάσταση de facto. Δεν υπάρχει. Συνεπώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε να το αφαιρέσει αυτό από τη ρητορική της. Δεύτερον, δεν λέει απόφαση τίποτα για τα ωφέλη του τοπικού πληθυσμού. Μιλάει για την συνένεση των Σαχαροή και το λέει αυτό ξεκάθαρα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν να διορθώσει παρακαλώ. Χρειάζεται συνένεση. Άρα με ποιον πρέπει να μιλήσουμε με το Πολυσάριο προκειμένου να υπάρξει εμπορική συμφωνία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν θα πρέπει να φροντίσει να υπάρξει συνάντηση με το Πολυσάριο για σχετικές συμφωνίες. Έπειτα πριν από λίγο πήραμε μια απάντηση ε, για το Κιμπέ. Από την Ισπανία την πήραν απάντηση. Πρόκειται για ένα αλλιευτικό σκάφος που έπρεπε να φανεί κατά πόσο ερχόταν από Δυτική Σαχάρα ή όχι το εμπόρευμα. Και λέει η Ισπανική κυβέρνηση ότι έχουμε δίκιο και ότι πρέπει να εφαρμόζεται η απόφαση του ΔΕΚ την πληροφορία αυτή την έδωσαν στη Γαλλία, η Γαλλία δεν ανταποκρίθηκε και είναι αλήθεια ότι δεν μπορούμε έτσι όπως έχουν σήμερα τα πράγματα να εφαρμόσουμε προνομιακή μεταχείριση στη Δυτική Σαχάρα. Και ρωτάω την Επιτροπή, τι θα κάνει για να βοηθήσει τις χώρες μέλη να σεβαστούν την απόφαση του δικαστηρίου. Πώς θα βοηθήσετε την Ισπανία για να μπορεί να ελέγχει από τη θάλασσα, από τον αέρα, ή οδικό τα εμπορεύματα τα οποία φτάνουν στη χώρα για να είμαστε σίγουροι ότι δεν είναι από τη Δυτική Σαχάρα. Και θέλω επίση να γνωρίζω ποιο είναι ο όγκο των προϊόντων που φτάνουν από τη Δυτική Σαχάρα και για πόσα χρήματα μιλάμε τα τελευταία δέκα χρόνια που δεν εφαρμόζουμε την ισχύουσα νομοθεσία. Ευχαριστώ. So, lot, Ευχαριστώ πολύ, συνάδελφοι. Να δώσω το λόγο τώρα στην Υπηρεσία εξωτερική Δράσης και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. τρει ομιλητέ τρία λεπτά έκαστος. Ο κ. Πικέ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σα είμαι ευγνώμων για τα σχόλια. Όσον αφορά την προσέγγιση μας. Θέλουμε να εφαρμόσουμε την απόφαση του δικαστηρίου δηλαδή τη νομική βάση για τις προτιμήσεις για τα προϊόντα με προέλευση Δυτική Σαχάρα. Αυτό γίνεται μέσω επίσημης τροποποίησης της συμφωνίας. Ακολουθώντας την κανονική διαδικασία της συνθήκης άρθρο 218 για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο θα εμπλακούν στη διαδικασία, όπως για οποιαδήποτε συμφωνία το δικαστήριο αναφέρεται στο ότι πρέπει να ληφθούν διάφορες στοιχές υπόψη για να προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρώτα απ' όλα χρειάζεται διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους λαούς. Να ληφθεί υπόψη το συμφέρον των λαών αυτών και η βιωσιμότητα. Είναι περίπλοκα θέματα. Χρειαζόμαστε λεπτομέρειες. Πρέπει να συζητηθούν με τους ομολόγους μας, με τους εταίρους μας. Το παίρνουμε πολύ σε σοβαρά το θέμα αυτό. Διότι θα καθορίσει την πολιτική και νομική ισχύ της προσεγγίσεώς μας. Θέλουμε να ακολουθήσουμε μια προσέγγιση που είναι βιώσιμη πολιτικός και προασπίσιμη. και ταυτόχρονα ε, συμμορφώνεται πλήρως με τις νομικές επιταγές. Αλλάζουμε τη Συμφωνία Σύνδεσης επίσης Ίσως, αλλά όχι τώρα. Πρέπει να περιμένουμε μέχρι να έχουμε σχετική απόφαση του ΔΕΚ για αυτή την συμφωνία. Και το ίδιο για την αλληλευτική συμφωνία. Οι αποφάσει αυτέ αναμένονται ίσως φέτος, ίσως και του χρόνου. Με αυτή την εκκρεμότητα δεν μπορούμε να φυσικάζουμε. Πρέπει να κινηθούμε τώρα όσον αφορά τη γεωργική συμφωνία. Δοθήσει της ε, επίπτωσης που έχει για το εμπόριο τώρα αυτή η συμφωνία. Ανέφεραν τα μέλη παραλληλισμούς Ουκρανία, Μολδαβία κλπ. Αυτή η περίπτωση πιστεύουν είναι αρκετά μοναδική για αντικειμενικούς λόγους. Ένα σημαντικότατος λόγος είναι και ο εξής. Για τη Δυτική Σαχάρα έχει κινητοποιηθεί η ειρηνευτική διαδικασία του ΙΕ. Θεωρείται μια αυτοκυβερνούμενη οντότης η Δυτική Σαχάρα πλευρά ΟΗΕ. Άρα αυτό διαφοροποιεί αυτή την υπόθεση από τις δύο αναφερθήσεις. Με ποιον έρχομαι σε επαφή, ποιος μας συμβουλεύει. πρέπει να το συζητήσουμε λεπτομέρως. Το δικαστήριο δεν αποφαίνεται επακριβώς όσον αφορά την προσέγγιση. Παραμένει ανοιχτό. Λέγει ότι απαιτούνται διαβουλεύσεις. Ποια η θέση του Πολυσάριο δεν καθορίζεται από το δικαστήριο που δεν είναι. Το Πολυσάριο πολιτικός αναγνωρίζεται ως εταίρος και εκπρόσωπος στα πλαίσια της ειρηνευτικής διαδικασίας του ΟΗΕ. Τίποτα άλλο. ότι πρέπει να επιληθεί προς όφελος των διμερών σχέσεων. Βεβαίως. Προφανώς δεν μπορούμε να αναζωογονήσουμε αυτή τη σχέση αν δεν βρούμε μία λύση. Δεν μπορούμε να πετύχουμε λύση για την σταθερότητα της περιοχής χωρίς να βρούμε λύση για το συγκεκριμένο. Ευχαριστώ κύριε Πιχέ. Κύριε Τζόστ, θα είμαι πολύ σύντομος, Πρόεδρε, λίγα λόγια για τα ήθη των προϊόντων που καλύπτονται από τη Γεωργική Συμφωνία. Τα προϊόντα είναι φωσφορούχα κυρίως από Δυτική Σαχάρα, κατεργασμένα ψάρια και ντομάτες. Ποια είναι η ιδέα. Όταν εξετάσουμε τις τροπολογίες των πρωτοκόλων, τις τροποποίησεις των πρωτοκόλων για να λύσουμε το θέμα της Δυτικής Σαχάρας και των σχετικών προϊόντων, δεν θέλουμε να ξεκινήσουμε μια συζήτηση για το μέγεθος των παραχωρήσεων. Οι παραχωρήσεις όσοι έχουν συμφωνηθεί με το Μαρόκο θα παραμείνουν. Πρέπει να διευκονίσουμε το θέμα της Δυτικής Σαχάρας. Άρα δεν θα επηρεαστούν οι ντομάτες. Οι περισσότερες ντομάτες δεν προέρχονται από τη Δυτική Σαχάρα, αλλά από το Μαρόκο αυτό κάθε αυτό και υπάρχει ένα σύστημα που μας επιτρέπει να χειριζόμαστε αρκετά καλά τις εισαγωγές του προϊόντος. Ευχαριστώ. Ο κ. Καστριγιαννάκης έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σε αυτή τη φάση ποια είναι η κατάσταση. Τα τελωνία δεν μπορούν να δεχτούν εισαγωγές προελεύσεως Δυτικής Σαχάρας. Δεν μπορούν να τύχουν αυτά τα προϊόντα προτιμησιακής ε, μεταχειρήσεως δεν αποτελεί απαγόρευση εισαγωγών, το επαναλαμβάνω. Δεν είναι θέμα παράνομης διακίνησης αγαθών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είναι θέμα του κατά πόσο εφαρμόζουμε ή όχι την προτιμησιακή προσέγγιση. Φυτογειονομικές συνθήκες πρέπει να εφαρμόζονται και για τα γεωργικά προϊόντα. Αυτό ξυπακούεται. Το θέμα για τα τελωνία είναι πώς να εντοπίσουν ενδεχομένως ενδεχόμενες εισαγωγές που θα ε, απαιτούν, θα θέλουν να τύχουν προτιμησιακής αντιμετώπισης και συνεργαζόμαστε με τις ελληνικές αρχές των κρατών μελών για να τις ευαισθητοποιήσουμε για το πρόβλημα. Νομίζω ότι είναι πολύ ευαισθητοποιημένες οι ελληνικές αρχές και να λάβουν τα αναγκαία μέτρα. Η συνεργασία όμως με το Μαρόκο, τα τελωνία του Μαρόκου είναι θεμελιώδου σημασία αν θέλουμε να βρούμε απαντήσεις στα ερωτήματά μας και να αποφύγουμε ε, διαταραχή όσον αφορά το εμπόριο. Αυτό είναι ένα θέμα που θα πρέπει να το συζητήσουμε στους συναδέλφους του Μαρόκου. Να προσθέσω και το θέμα της ετικητοθεσίας ακολουθεί άλλη νομοθεσία. Δεν σχετίζεται με το κατά πόσο θα εφαρμοστούν προτιμησιακά μέτρα σε αυτό το εμπόριο. Ευχαριστώ. Ίσως επικρατεί μεγαλύτερη σαφάνεια, δεν έχει βρεθεί λύση. Οπότε θα συνεχιστεί η συζήτηση, όμως θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους και τους εκπροσώπους της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα σχόλιά τους. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης την ΑΦΕΤ για την θαυμάσια συνεργασία σας μαζί μας και καλή συνέχεια της συνεδρίασης. Ευχαριστώ αγαπητέ Λάγκε. Αποχαιρετούμε τους συναδελφούς μας της Επιτροπής ΙΝΤΑ, Διεθνούς Εμπορίου. Θα συνεχίσουμε βέβαια τη σκληρή εργασία μας εμείς της Επιτροπής Εξωτερικών. Διακόπτει ο Πρόεδρος. the... Βεβαίως ε, οι μισοί φαίνεται πως έχουν πάρει μεταγραφή στην ε, Επιτροπή Εξωτερικών, στην Επιτροπή μάλλον ε, Διεθνούς Εμπορίου. Αν θέλετε να αποχωρήσετε από την αίθουσα να το κάνετε, αλλά εμείς εδώ έχουμε πολλή δουλειά ως Επιτροπή Εξωτερικών και δεν μπορούμε να περιμένουμε. Σας παρακαλώ λοιπόν